Please take your seats. We want to start. Please, please take your seat. We want to start. Please. Παρακαλώ καθίστε να ξεκινήσουμε. Se siamo pronti a cominciare, prego. Αν είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε, παρακαλώ καθίστε. Προτείνω, αν συμφωνείτε, να κάνουμε μια επαλήθευση με την ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά αποχές. Άρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει, άρχισε η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πέρας. Ξαναρχίζουμε την ψηφοφορία. Ας ψηφίσουν όλοι παρακαλώ. Πέρας. Ε, επαλήθευση, επαλήθευση. Ας προχωρήσουμε λοιπόν αμέσως στην ψηφοφορία μας και μετά θα αναλάβει ο συνάδελφος Φέντερλε την προεδρία στη συζήτηση. Όχι. Πρόεδρε, ναι, ευχαριστώ. Ο κύριος Σαφοζέχ. Μια και η έκθεσή μου αναδιατυπώθηκε μέσω των τροπολογιών που την τροποποίησαν τόσο πολύ, δεν την ψηφίζω. Εφόσον περάσουν οι τροπολογίες αυτές. Δεν την υπερψηφίζω και παρακαλώ να αποσυρθεί και το όνομά μου. Και ευχαριστώ. Εντάξει, τα ακούσατε όλοι. Βεβαίως και καταγράφουμε αυτήν σας τη δήλωση και μετά την ψηφοφορία βλέπουμε αν θα προχωρήσετε στην αποχώρηση. Κύριε Σαφοζέχ, και έχουμε ένα κατάλογο αρκετά μακροσκελή αλλά και ψηφοφορίες σαν μπλοκ. Οπότε μπορούμε να πάμε σχετικά σύντομα ε, με την τροπολογία 63 πρώτα και 64 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65-66 καταπίπτουν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι νωρίς ξέρω, αλλά κάντε μια προσπάθεια να σηκώνετε το χέρι σας και όχι μόνο συντονιστές. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 71 υπέρ κατά αποχές σαν να εγκρίνεται εγκρίθηκε 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, καλά, μη φωνάστε, σας ζητήστε μια επαλήθευση και να το κάνουμε. Αμέσω. Άρχεται η ηλεκτρονική επαλήθευση. 73 της κυρίας Ματίας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και απερίφθη. Και μάλιστα με το παραπάνω. Λοιπόν, 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 75. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται. Και θεωρώ ότι έχει εγκριθεί. Ας δούμε τι μας λέει και το σύστημα. Ενεκρίθη. 76 δύο τμήματα υπέρ στο πρώτο παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές και παληθεύουμε ηλεκτρονικά για να βεβαιωθούμε. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν της τροπολογίας 76 πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές και απερίφθη. 79 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 3 ύμκο. Ποιος θέλει παλήθευση. Στην 85 η Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τρία της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86, 87 και 88 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 90 και 89 καταπίπτουν, 92 τώρα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 93-94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95-96-97 κατά πίπτου 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, unblock η 100 και 101 Α, πάω πολύ γρήγορα, μα γιατί. 100 και 101 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 102 καταπίπτει, 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 105 103 υπέρ αποχές εγκρίνεται. Θέλετε παλήθευση. 105 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Unblock από την 106 ως την 116 συμπεριλαμβανόμενοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ήμκο 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117-118 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 119 και 120 καταπίπτουν 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ Πέρασε. Απερίφθη. 123, 24, 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 126 καταπίπτει 128 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 127, 128, 129 130 υπέρ κατά. 130, 131, 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 134, 135, 136 block υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139, 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141, 142, 143 unblock υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 146 έως και 152 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 146 και ΙΜΚΟ 7 on block υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 153, 154, 155 on block, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, καταπίπτει 156, 157, 159, 161, 162 ομού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 158 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 160 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Λίμπε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 της Λίμπε υπέρ κατά αποχές μάλλον απερίφθη. 164-165 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν μάλλον αν δεν ζητάει κανείς επαλήθευση 166 καταπίπτει ε, όχι, πρέπει να την ψηφίσουμε. «166, 167, 168, 169, ομού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 170 κατά πίπτη, 171 έως και 176 ομού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178, 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 κατά πίπτη, 182 186. Τέσσερις τροπολογίες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 8 τη ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 τη ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται 181 υπέρ κατά εγκρίνεται 183 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 187 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 σε 191 on block υπερκατάποχες αποχές εγκρίνονται. 192 καταπίπτει, 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Οι 194 και οι 5 και 6, 3 ε, ε, υπέρ κατά ε, εγκρίνονται, 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 198 υπέρ κατά εγκρίνεται, καταπίπτουν οι 199 και οι 200, 201 υπέρ κατά εγκρίνεται. 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 203, 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 205 και 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Καταπίπτουν 207 και 8. 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 έως και 14. Οι 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 216, 17 και 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Καταπίπτουν οι 219 και 220 από την 221 μέχρι και την 223. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Κατά πίπη 224. 225 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 220 ήταν 226 πριν, 227 τώρα. Εγκρίνεται 227, 228 και 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 231, 32 και οι δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 233 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 234 έως και 236 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 237 καταπίπτει, 238 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 240, 41 και 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 243 καταπίπτει, όλες μαζί, 244 μέχρι και την 251 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Λίμπε, 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε, 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμκο, 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 252, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 253 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 254 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 250 θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 254 Α, του Ashley Fox έναρξη ψηφοφορίας ψηφίζουμε τώρα come, come, Άρα απορρίπτεται, εντάξει. 255 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 256 υπέρ κατά αποχές. Α, και εδώ θα πρέπει να γίνει επαλέψη νομίζω απορρίπτεται. Για το 256 ψηφίζουμε τώρα. Ψηφίζουμε πέρας και εγκρίνεται. Άρα ορθώς κάνουμε την επαλήθευση, έκανα λάθος. 2.57 υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 2.58 εγκρίθηκε το 57. 2.58 υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 2.59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 260 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 έως και 4. Κατά αποχές εγκρίνονται. 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από το 6 μέχρι και το 15. Όλες μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 7. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10. Για το 9 θέλετε έλεγχο. Είμαι σίγουρη ότι απορρι... απορρίφθηκε. Για το 10. Για το 10 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας κάνουμε έλεγχο για το 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται από το 17 μέχρι και το 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται από το 20 μέχρι και το 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 μέχρι και το 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 μέχρι και το 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 34 υπέρ. 34 επαναλαμβάνει η πρόεδρος. Εγκρίθηκαν οι προηγούμενες. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από το 35 μέχρι και το 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από το 39 μέχρι και το 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 έως και 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από το 47 μέχρι και το 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51, 52 και 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Καταπίπτει το 54, 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 και 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Καταπίπτουν το 58 και το 59 και ψηφίζουμε το 60 μέχρι και το 62. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Λίμπε α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία. Και αυτό το οποίο πρότεινε ο κ. για την απόσταση του νόμου του εφόσον πέρασαν οι τροπολογίες, νομίζω ότι θα πρέπει να αποσύρουμε το όνομά του τώρα από την έκθεση, άρα να συμφωνήσουμε με την πρότασή του. Νομίζω ότι έχουμε τώρα έγκριση αυτής της ε, έκθεσης που θα κατέβει στην Ολομέλεια χωρίς το όνομα του εισηγητή. Τελική ψηφοφορία. Τώρα ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με 47 ψήφους υπέρ. Ευχαριστούμε και Σοφάζο που διευκολύνατε την ολοκλήρωση της διαδρομής του θέματος και που θα κατέβει στην Ολομέλεια. Και τώρα θα συνεχίσει στην Προεδρία ο συνάδελφος Φέντερλε. Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Ήταν ε, μια πολύ ομαλή ε, και γρήγορη ε, ψηφοφορία. Ήταν λίγο δύσκολο να την παρακολουθήσει κανεί μερικέ στιγμέ, αλλά εν πάση περιπτώσει εξοικονομήσαμε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πολύ που μου επιτρέπετε να αναλάβω την Προεδρία για το τελευταίο τμήμα τη συνεδρία. Να αρχίσουμε με την έγκριση ημερήσια διάταξη. Θέλει κανεί να πάρει το λόγο βλέπω ότι δεν υπάρχουν σχόλια, άρα εγκρίνεται η μισή διάταξη. Θα ήθελα να σας πω στις ανακοινώσεις του Προέδρου το σημείο 8 ε, ο κύριος Κένκελ έχει ζητήσει αν είναι δυνατόν ε, τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το σχέδιο γνωμοδότησή του, να ε, συζητηθεί στις 6 Φεβρουαρίου. Αναβάλλεται λοιπόν για σήμερα. Πάμε στο σημείο 3, που είναι η έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 26 Σεπτεμβρίου 12 και 13 Οκτωβρίου 16 και 9 με 10 Νοεμβρίου του 2016. Υπάρχουν, υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά. Αν όχι, θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά αυτά. Περνάμε τώρα στην έκθεση για το σχέδιο δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016 με 2020. Η Αγγέλικα Μίναρ είναι ε, η συντάκτη γνωμοδότησης. Ε, υπήρξε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020. Η ΙΜΚΟ είναι η επί τη ουσία αρμόδια, Όμω εμεί υπό τον κανόνα 54 συμμετέχουμε. Έχουμε ειδικέ αρμοδιότητε λοιπόν για ορισμένα τμήματα της ε, έκθεσης. Ε, σήμερα εξετάζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ε, της κυρίας Μιλίναρ. 40 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Πρώτα θα μιλήσουν οι συγητές, μετά οι σκιώδεις συγητές και μετά θα δώσουμε τη δυνατότητα για ένα λεπτό σε όλους τους συναδέλφους που το επιθυμούν να πάρουν το λόγο και μετά θα συνοψίσουν μα συνοψίσει η εισηγήτρια, η συντάκτα τη νομοδότηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ανάπτυξη τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι βασικό τμήμα τη ε, στρατηγική για την ψηφιακή αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση τη αποδοτικότητα, τη μείωση ε, του κόστου και τη μείωση τη γραφειοκρατία ε, προ όφελο των πολιτών. Οπότε, εγώ επικροτώ την το σχέδιο δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2016 μέχρι το 2020. Υπάρχουν σημεία που είναι ε, ιδιαίτερο ενδιαφέροντο για την Επιτροπή μα. Έχουμε αποκλειστική είτε ε, κοινή αρμοδιότητα με την ΙΜΚΟ υπό τον κανόνα 54. Ένα βασικό σημείο είναι ότι πρέπει να υπάρξει μακροπρόθεσμη ε, ένα μακροπρόθεσμο βιώσιμο πλαίσιο ε, και μετά το 2020. Πρέπει να εξασφαλίσουμε συγκεκριμένα τη βιωσιμότητα όλων των ήδη δρομολογηθέντων ε, προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα την διευκόλυνση για τη σύνδεση της Ευρώπης, μεταξύ άλλων. Πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα, να είναι φιλική προς το χρήστη η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, γιατί οι υπηρεσίες είναι πάρα πολύ βασικές. Έχουμε ραγδαία αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, ε, το διαδίκτυο των πραγμάτων, το υπολογιστικό νέφος, όλα αυτά που μεταλάβουμε να υπόψη καλύτερα ως προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προκειμένου οι υπηρεσίες ε, να μπορούν να ανταποκριθούν στην πρόκληση τη εξέλιξη τη τεχνολογία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τι καλύτερε υπηρεσίε στο πλαίσιο τη ηλεκτρονική ε, ε, διακυβέρνηση. Πρέπει οι υπηρεσίε και τα δεδομένα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ε, Επομένω, η συμπράξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικό παράγων για τι νέε καινοτόμε λύσει που θα προκύψουν. Δεν πρέπει να ξεχνούμε όμω ότι για να ε, ε, λάβει, να ληφθεί υπόψη και το μέλλον, πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη κάποια στοιχεία, κάποιες υποδομές ε, ε, όπως για παράδειγμα η ζωνική ε, πρόσβαση και η χρήση ραδιοσυχνοτήτων ειδικότερα για την, για τις, για την τηλεφωνία, η αξιοποίηση όλης αυτής της προσπάθειας είναι πολύ χαμηλή σε ορισμένες, κάποια, σε ορισμένες χώρες. Είναι λοιπόν σημαντικό να, είμαστε πιο, να είναι όλα αυτά περισσότερο προσαρμοσμένα σε σχέση με τις ε, ανάγκες των χρηστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πρωτοστατήσει μέσω του παραδείγματός της. Επομένως, ε, θα θέλαμε να προωθήσουμε την περαιτέρω ψευιοποίηση των ε, ευρωπαϊκών θεσμών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να πρωτοστατεί ακόμα περισσότερο στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οπότε εγώ με χαρά ε, περιμένω τις ε, τροπολογίες των συναδέλφων, μας, ε, των συναδέλφων μου και την συζήτηση που θα γίνει κατά τις ερχόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μλίνα. Περνάμε στους κοιόδης εισηγητές. ΕΛΚ. Κυρία Σάντερ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αγγέλικα Μινάρ για την εξαιρετική εργασία που μας προτείνει σήμερα. Η δική μου συνεισφορά ε, αφορά την προστίκη κάποιων ιδεών ε, επειδή έχουμε περιορισμό στον αριθμό ε, χαρακτήρων, δεν μπόρεσε να τα συμπεριλάβει. Αναφερθήκατε στην ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών που είναι επικερδής για όλους ως προς το κόστος ως προς την αποδοτικότητα και ως προς τη διαφάνεια και επίσης ε, μειώνεται η γραφειοκρατία ε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις μας ε, και κυρίως για τις μικρομεσαίες. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι <clears throat> η αρχή only ε, once, άπαξ μόνο, αν, θα μπορούσαμε, να την ε, εφαρμόσουμε, 5 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' ε, Και ένα σημείο που θα ήθελα επίσης να τονίσω είναι να σας, να σας υπενθυμίσω ότι βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι η εμπιστοσύνη, επομένως η ασφάλεια των υποδομών είναι πολύ σημαντική. Δεύτερο πολύ σημαντικό είναι η ψηφιακή ένταξη. Ε, δεν πρέπει να ε, γίνει ε, πλήρως, ε, να υπάρξει πλήρης ψηφιοποίηση. Πρέπει να ληφθούν υπόψη μερικές ευαίσθητες ομάδες, όπως για παράδειγμα άτομα με αναπηρίες ή ηλικιωμένοι, που δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες της ψηφιακής, επομένως πρέπει η διοίκηση να παραμείνει παρούσα για να μην υπάρξει ψηφιακό χάσμα. Όσον αφορά τις μεθοριακές περιοχές μας, θα θέλω να επιμείνω στη συνέχεια των δημοσίων υπηρεσιών διασυνοριακά και την συνεργασία των διοικήσεων διασυνοριακά, Οπότε ελπίζω ότι σύντομα θα υπάρξει ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με την κοινωνική ασφάλεια ε, όπως ε, επίσης να επιμείνω στη σημασία του να είναι κατανοητές ε, και εύχριστες η χρήση, η χρήση, η χρήση των ε, ε, ψηφιακών υπηρεσιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, σκιώδης εισηγητής των φιλελευθέρων. Κύριος Ζωρίνιο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή της δουλειά. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, βήμα ε, της ε, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα αυτό διευκολύνει την διαλειτουργικότητα. Υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές που αναφέρονται, τονίζονται ιδιαίτερως το Κοινοβούλιο ε, πρέπει να επιμείνει στην ε, ύπαρξη μιας ε, ευρωπαϊκής πλατφόρμας αναφοράς για την για τη διαλειτουργικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι η βάση, αλλά αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο δράσης για την ύπαρξη και την εφαρμογή αυτής της πλατφόρμας, ε, δεν θα μας είναι ποτέ χρήσιμο στην πράξη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ορίσουμε τις προτεραιότητες όσων επιθυμούμε να κάνουμε στο πλαίσιο αυτής της πλατφόρμας και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ε, τροποποιήσουμε το σχέδιο δράσης, ε, το, συγγνώμη, την, ε, το σχέδιο γνωμοδότησης. Έχουμε βέβαια περιορισμό χαρακτήρων, πρέπει όμως να ενισχύσουμε την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία της αύξησης ποιότητας των ε, υπηρεσιών που παρέχονται στο πολίτη, να είναι ε, εστιασμένοι περισσότεροι στις ανάγκες ε, των πολιτών και όχι μόνο στις πτυχές τις καθαρά ψηφιακές ή στα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Υπάρχει λοιπόν, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανάγκες των χρηστών Λοιπόν, με την, σε συνδυασμό με την, την αύξηση των θέσεων απασχόλησης ε, ε, πρέπει λοιπόν ε, να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις ανάγκες των χρηστών και όχι τόσο στα επιχειρηματικά συμφέροντα και στις τεχνικές, τεχνολογικές πτυχές. Πρέπει ο κόσμος να έχει στη διάθεσή του πιο εύχριστες υπηρεσίες και στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου δράσης ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συμπεριβαλάβουμε και ένα πακέτο για τις ε, τηλεπικοινωνίες με τέσσερις ε, τομείς, για παράδειγμα το 5G, ε, την πρωτοβουλία ε, Wi-Fi για την Ευρώπη, για την οποία εγώ είμαι εισηγητής, ε, να υπάρξουν οι συνθήκες συμμετοχής και πρόσβασης σε ένα σε ένα ίντερνετ, σε ένα διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας. Δεν έχουμε και τόσο πολύ χρόνο, οπότε θα πρέπει ο κάθε ένας από εμά ε, να περιορίζεται ε, στο χρόνο του για να μπορέσουμε να ε, μην καθυστερήσουμε. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Οι σκιώδεις ηγητές των Πρασίνων και των Συντηρητικών δεν εδώ. Πάμε τώρα στην κυρία Ματιάς λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Νομίζω ότι αυτό το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πολύ ε, σημαντικό για διάφορους λόγους. Ε, δεν χρειάζεται δύο φορές ε, να εκδίδεται το ίδιο έγγραφο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και από γραφειοκρατικής απόψεως. Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να είμαστε πιο περιεκτικοί στην προσέγγισή μας. Καταλαβαίνω ότι έχουμε περιορισμό στον αριθμό χαρακτήρων, δεν είναι δυνατόν να τα καλύψει κανείς όλα. Το γνωρίζω αυτό πολύ καλά. Όμως νομίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να προσθέσουμε, να ενισχύσουμε δύο στοιχεία τα οποία σε κάποιο βαθμό αναφέρονται έμεσα, όμως πιστεύω ότι πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω σχέδιο δράσης λοιπόν πιο αποτελεσματικό και ε, πιο περιεκτικό ε, παρά τις ε, νέες τεχνολογίες που τα πηγαίνουν πολύ καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόσβαση όμως είναι πολύ άνηση και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με αυτήν την ανισότητα πρόσβασης. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι έχουν μία πραγματική πρόσβαση στο δίκτυο αυτό. Δεύτερον, προστασία των δεδομένων, ασφάλεια των δεδομένων, επίσης πρέπει να αναφερθεί. Αναφέρεται ε, από την εισηγήτρια, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναπτυχθεί. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε η ε, νομοθεσία όσον αφορά την προστασία ε, δεδομένων, που είναι μια πολύ καλή νομική βάση, να εφαρμόζεται πραγματικά. Και τελευταία παρατήρηση, διαφωνώ με ε, ένα θέμα και θα υποβάλω και τροπολογίες ε, σχετικά η συμμετοχή των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού ε, τομέα. Νομίζω ότι τα επιχειρηματικά συμφέροντα δεν πρέπει να κερδίζουν έναντι των συμφερόντων των πολιτών και πρέπει να δοθεί λιγότερη σημασία κατά τη γνώμη μου στο ρόλο που διαδραματίζουν οι συμπράξεις αυτές πρέπει να αναφερθούμε περισσότερο στις συμβουλευτικές υπηρεσίες ε, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και στις επόμενες συνεδριάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ματιάς. Ο κύριος ε, Λόπετ από τους ε, Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα αυτός ο μεγάλος μετασχηματισμός, η αλλαγή που έχει σχέση με τις νέες τεχνολογίες ε, επιβάλλει το να πώς αρμοστούμε στους νέους καιρούς, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να μειώσουμε τις ε, δαπάνες, τις δαπάνες τις διοικητικές. Αυτό όλα θα έχουν πάρα πολύ ευεργετικές συνέπειες για τις ε, επιχειρήσεις. Περικοπή το δαπανών σημαίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Όπως αναφέρθηκε, έχουμε νέες ευκαιρίες αλλά και, και νέους κινδύνους. Τελικά είναι θέμα προστασία των δεδομένων, οπότε και επισύρω την προσοχή σας στο εξής. Η τεχνολογική πρόοδος δεν θα πρέπει στο να διευρύνει, να μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ εκείνων που έχουν πιο εύκολη προσβασιμότητα στις νέες τεχνολογίες ε, σε σχέση και με τα αντίστοιχα πρόσωπα και μεταξύ των άλλων. Άρα θα πρέπει να αποφύγουμε η πρόοδος τεχνολογίας να δημιουργεί χάσμα μεταξύ κατηγοριών πολιτών ή χωρών. Πρόεδρος. Δεν έχει ζητήσει άλλο συνάδελφο τον λόγο. Άρα πάμε στην Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Είναι Γιούνκερ από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Σας Ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε ξανά στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πρώτα πρώτα το Κοινοβούλιο αλλά και την ε, Επιτροπή Ήτρε. Όλα αυτά ε, είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τα όσα διαπιστώσαμε. Το πόσο η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει ε, την διοίκηση, τη διαχείριση, ε, για τη σχέση τέλος πάντων των φορέων αυτών με την ε, κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια εμείς να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Άρα θα πρέπει και τα άλλα θεσμικά όργανα ε, να κάνουν το ίδιο. Αυτά θα έχουν επιπτώσεις σημαντικές και θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι το νέο πρόγραμμα δρασίας το προηγούμενο έχει και μια δυναμική διάσταση δηλαδή αυτές οι δράσεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα θα συμπληρωθούν από άλλες δράσεις. Και συγκεκριμένα φτιάξαμε αυτή την πλατφόρμα. Εκεί να ακούσουμε τους εμπλεκόμενους, δηλαδή και επιχειρήσεις και πολίτες. Να δούμε και να επισημανθεί σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη ποιες είναι οι δράσεις, οι καινούργιε που πρέπει να γίνουν, ούτω ώστε τελικά την μεταμόρφωση, την αλλαγή στη δημόσια διοίκηση να την επιταχύνουμε γιατί περί αυτού πρόκειται. Πολύ θετικά ε, αυτά τα οποία άκουσα. Είναι θετικό που το συμμετέχουν και στη συζήτηση τη δική σας και σας ευχαριστούμε Πρόεδρος. Ευχαριστούμε εμείς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δηλώση τούτη. Και θα επανέλθουμε τώρα στην εισηγήτρια για να δευτερολογήσει και ολοκληρώσει. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους λέει η, εισηγήτρια. Ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν εδώ και νομίζω, λέει κυρία Μίλναρ, ότι εδώ μπορώ να ολοκληρώσω το ότι θα πρέπει να έχουμε τελικά μια γνωμοδότηση ε, αποκρισταλωμένη, κατασταλαγμένη και το μεσημέρι 17 Ιανουαρίου λίγη προθεσμία υποβολής των τροπολογιών στη συνέχεια. Βέβαια θα συνεχίσουμε τη διαδρομή αυτή ε, και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Ε, εμείς ευχαριστούμε Κύριε Μίλαν λέει ο πρόεδρος και εδώ ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση για το σχέδιο δράσης διακυβέρνησης 16-20. Σας ε, ανακοινώ ότι θα ψηφίσουμε στις 28 Φεβρουαρίου και ακόμη δεν έχει δηλωθεί το πώς θα γίνει ψηφοφορία στην Ελλομέλεια, αλλά τέλος πάντων πρέπει να σας πω ότι πάμε καλά με το χρονοδιάγραμμα Και θα πρέπει βέβαια να προλάβουν να έρθουν οι συνάδελφοι για τι επόμενε συζητήσει. Τώρα πάμε στο 7ο θέμα. Ετήσει μείωση εγωγών αερίων θερμοκηπίου ε, ε από το μέλλον 21 έω 30 για την Ενεργειακή Ένωση. Τον ε, Ιούλιο κατέβασε κάποια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έναν ε, κανονισμό. Και εκεί λέει για δεσμευτικέ προβλέψει και στόχου για τι εκπομπέ για την περίοδο 2021-2030 και πρόκειται για κάποιους ε, στόχους οι οποίοι καλύπτουν διάφορους τομείς ε, εκτός ε, του ETS και αυτό σημαίνει 60% του συνόλου των εκπομπών της Ένωσης. Έχουμε αυτή την πρόταση η οποία αποτελεί την συνέχεια στην effort sharing decision, στην απόφαση για την κοινή προσπάθεια σε σχέση με τους εθνικούς στόχους 2020. Ε, ε, η ΕΝΒΗ είναι η αρμόδια επιτροπή, κάναμε ανταλλαγή απόψεων το Νοέμβριο. Ε, προβλέπονται 30 λεπτά για αυτό το θέμα, να κάνουμε την κλασική διαδικασία, να ξεκινήσει ο εισηγητής, δεν είναι εδώ όμως, έρχεται από ό,τι μου είπαν. Α, νάτος, νάτος, ήρθε, ήρθε, ήρθε. Ωραία. Ένα λεπτάκι για να καθίσει και συνεχίζουμε. Πάντως, πάντως, κανείς αποδίδει καλύτερα στις ε, αγορεύσεις όταν έρχεται βιαστικά συνεδρίαση. Welcome. Έγινε γρήγορα ψηφοφορία και όλοι συμβάσκαν τα χρονικά όρια, γι' αυτό και ε, φτάσαμε πιο νωρίς σε αυτό το σημείο. Δεν φταίτε εσείς που περιστερήσαμε λίγο. Έχετε το λόγο κύριε Ιζήγητη. Στην ένβη είχα μια υποχρέωση πρόεδρε, γι' αυτό άργησα. Α, τελικά τα κατάφερα όμως. Για να δούμε. Όσον αφορά αυτόν τον κανονισμό της κοινή προσπάθειας, ε, είναι σημαντικό το θέμα γιατί καλύπτει το σύνολο των εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για βασικό μέσο καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, φαινόμενο που το ξέρουμε όλοι. Λέει το σχέδιο κανονισμού ότι θέλουμε νέα όρια και μείωση για την ε, περίοδο 2021 έως 30. Όσον αφορά τώρα το Κοινοβούλιο, γνωμοδοτούμε, η αρμόδια επιτροπή είναι η ΕΝΒΗ, εμείς έχουμε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους εκείνης της επιτροπής. Ο κύριος Χερμπράντι είναι ο εισηγητής. Βεβαίως και έχουμε αποκλίνουσες απόψεις εμείς από εκείνους αλλά προσπαθούμε να έχουμε κάποια συνέπεια στα όσα λέει το κείμενο του καθενός. Χθε είχαμε μια τυπή συνεδρία των ε, συντονιστών και των εισηγητών και από τις δύο επιτροπές από πολιτικά κόμματα. Νομίζω ότι επεδείχθη καλή πίστη, καλή διάθεση από όλους τους κοιοδεσηγητές και θεωρώ ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να επιληθούν. Και ακριβώς με τη στενή συνεργασία των σκιωδών θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση η οποία να είναι ικανοποιητική για τις πολιτικές ομάδες και τους συναδέλφους. Έχουμε πέντε σημαντικά σημεία. Πιστεύω ότι επ' αυτών θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Πρώτον, αύξηση ε, των όσων προβλέπουμε, δηλαδή να ανέβει ο πύχης. Έχουμε δεδομένη τη Συμφωνία των Παρισίων, έχουμε επίσης τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις της Ένωσης που αφορούν τον άνθρακα. Δεύτερο σημείο είναι το πότε θα έχουμε την αφετηρία, πού θα έχει διαδρομή του αυτός ο κανονισμός, οπότε να μην έχουμε αχρίαστη αύξηση της προοικοδότησης και να έχουμε πιο αυστηρή ρύθμιση, ζητώ να έχουμε μια γραμμική διαδρομή, δηλαδή να ξεκινήσουμε το 17 και σε αυτό συμφωνία και η ένβη. Και από όσο διαπίστωσα χτες, συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες. Μετά, μηχανισμοί ευελιξίας. Εδώ είναι το πιο δύσκολο σημείο της έκθεσης. Να δούμε πώς θα χειριστούμε τον παραδοσιακό αλλά και τον νέο κανονισμό όπως προτείνει. Ε, πρέπει, πρέπει να ανακλείσεις ε, για βόρ, διότι τέλειωσε το τρίλεπτο. Επομένω, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον η συμμόρφωση, τι γίνεται και επίση και με την αξιολόγηση η αναθεώρηση του κανονισμού. Και νομίζω ότι από αυτού του σημείου θα πρέπει να γίνει πρόταση για πιο τακτικούς ελέγχου συμμόρφωσης των κρατών μελών και θα πρέπει όσο γίνεται πιο νωρίς να αφιερθεί ο κανονισμό για να είμαστε σίγουροι ότι όλα πάνε καλά. Για βόρεια συγγνώμη που σε ε, πίεζα, αλλά ε, ξέρετε, εμεί είμαστε πιο Γερμανοί από Γερμανούς Γερμανού ω Σουηδοί. Δηλαδή θέλουμε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Πράγμα το τύπο ότι έχουμε χρόνο. Τέλο πάντων, θα δούμε τώρα του αγορητέ των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Κέλλη για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή, αλλά και προς την Επιτροπή. Εύστοχα όσα λέει η Κομισιόν. Άρα, να ισχύσει η πρόταση της Κομισιόν. Ίσως πάει μακριά ο εισηγητής. Και αυτό θα έχει επιπτώσεις όσον αφορά τη σχέση κόστους, αποτελέσματος, όσον αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία, όσον αφορά την απασχόληση, αλλά και την ασφάλεια. Τη διατροφή. Τέλος πάντων, όλοι συμφωνούμε για τον στόχο του 2030. Για τον στόχο συμφωνούμε, αλλά για τα μέσα επίτευξης όχι. Άρα, θα πρέπει να συμμορφωθούμε πρώτα-πρώτα με τη Συμφωνία Μαρακές και με την ε, Συμφωνία των Παρισίων. Εγώ ε, προσώπησα το Κοινοβούλιο και στις δύο αυτές συναντήσεις. Άρα, ποια θα πρέπει να είναι η αφετηρία. Το 2020 είναι εύστοχη επιλογή από την Επιτροπή. Ο συγκεκριτής λέει 2017. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι πολύ νωρί. Έτσι θα δυσκολευτούν τα κράτη-μέλη. Ε, ίσως δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί. Οπότε θα υπάρξουν συνέπειες. Δεύτερον, αναφέρθηκε ο συγκεκριτής ε, μέσα ευελιξίας και εν προκειμένου νομίζω ότι καλά τα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που λέει ο νομίζω θα έχει επιζήμια αποτελέσματα. Αυτές οι περικοπές είναι και θέμα διατροφικής ασφάλειας του, που είναι ε, κάτι το βασικό που προβλέπεται σύμφωνα των Παρασιών επίσης και για την ευελιξία του συστήματος προστόσεων του ETS θέλει να κατέβουμε στα 50 ο εισηγητής 100 ε, όταν υπάρχει εξοικονόμηση εκπομπών είναι δεδομένο αυτό και εδώ θα πρέπει να προλάβουμε τις εξελίξεις, τις σημαντικές όπως το Brexit. Άρα, να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Πάντως ευχαριστούμε και εισηγητή και την Επιτροπή. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Α, τα πήγατε πολύ καλά. Να πώς μπορεί κανείς να τηρήσει το χρονικό πλαίσιο. Πάμε τώρα στους σοσιαλιστές. Κύριε Μποναφέ. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω και εγώ την ίδια στρατηγική, πας και κερδίσουμε λίγο χρόνο. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης και για τη συνάντηση που είχαμε χτες. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση, η οποία θα συμπληρώσει τη στρατηγική για να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας από τη διάσκεψη των Παρισίων και να εξασφαλίσουμε ένα οικονομικά βιώσιμο μοντέλο χαμηλών εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Στην Επιτροπή ΕΝΒΙ είχαμε το ETS αυτή την εβδομάδα και βέβαια και ε, τους λοιπούς τομείς τους λέγουμε σε αυτή την έκθεση. Από το 2020 στο 2030 λοιπόν θα έχουμε χρόνια κρίσιμα για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναλάβαμε. Η πρόταση της Επιτροπής είναι και για μένα ένα καλό σημείο κίνησης. Οφείλω να πω ωστόσο ότι σε κάποια σημεία θα πρέπει να αναλάβουμε οπωσδήποτε δράση. Πρόκειται για τα σημεία που ήδη επεσήμαναν οι συνάδελφοι και κυρίως η συγγήτρια, για ο εισηγητής, ιδιαίτερα για τις προδιαγραφές που προβλέπονται και την αναθεώρηση, επαλήθευση και ενδεχόμενη αναθεώρηση των νέων πιλωτών για ευελιξία και στο σύστημα ITS και στο USF ε, πρέπει να το πράξουμε αυτό με βάση και τα όσα θα προκύψουν ε, στις σχετικές εργασίες του Κοινοβουλίου. Σημείο κίνηση λοιπόν ε, για την πορεία μείωσης των εκπομπών. Το σύστημα προχωράει, θα χρειαστεί οπωσδήποτε αναθεώρηση διότι δίνει αυτή τη στιγμή πλεονέκτημα σε όποιους έχουν καθυστερήσει στην καινοτομία, δεν έχουν κάνει επαρκείς πρόοδους και έτσι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση οι χώρες που έχουν προχωρήσει προς στην επέτευξη των στόχων. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και το σύστημα επαλήθευσης των, της των στόχων με αιτήσει εκθέσεις που θεωρούμε πολύ σημαντικές και πρέπει βέβαια να βελτιωθεί η επαλήθευση σε πενταετή βάση. Όπω είπαμε λοιπόν, καλές οι προθέσεις, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε προτάσεις για να βελτιώσουμε και να έχουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Επί τη ουσία, ευχαριστώ πολύ. Εκπρόσωπο του ECR δεν βλέπω. Άλτε. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Κύριε Βίνη. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, όπως είπατε, ε, μιλάω εκ μέρου ε, τη κοιόδουση ηγήτρια των Φιλελευθέρων που δεν μπορούσε να είναι εδώ. Η κυρία Πούντσετ θα ήθελε λοιπόν να ευχαριστήσει τον ε, εισηγητή για την προσπάθειά του. Θα ήθελε όμω να καταστεί το κείμενο πιο φιλόδοξο. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να ενισχύσει περισσότερο την μακροπρόθεσμη φιλοδοξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό το μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης ε, των εκπομπών αερίων ε, θερμοκηπίου. Πιστεύει ε, ότι είναι καλύτερα να αρχίσουμε το 2017 και όχι το 2020, γιατί το 2020 θα έχουν μειωθεί αποτελεσματικότερα οι εκπομπές και έτσι η πορεία θα είναι καλύτερη. Όσον αφορά τους μηχανισμούς ευελιξίας, η, η συγκήτρια πιστεύει ότι μπορεί να είναι σημαντικά εργαλεία για τα κράτη-μέλη, όμως πρέπει να, δείχνουν αποδεικνύουν ε, πραγματικά ωφέλη ως προς τη δυνατότητα των κρατών μελών να μειώσουν τις εκπομπές ε, αερίων θερμοκηπίου. Ειδικότερα όσον αφορά ε, τα 190 εκατομμύρια που θα δοθούν ε, όσον αφορά την ενίσχυση των δασών, ε, μεταξύ άλλων, ε, πρέπει να διατηρηθούν, όμως παράλληλα πρέπει να εγγυάται η επιβίωση, να εγγυόμαστε την επιβίωση του αγροτικού τομέα. Προτείνει αναθεώρηση κάθε πέντε χρόνια, ενώ ο εισηγητής προτείνει κάθε χρόνο. Ε, θα προτείνει όμως ένα συμβιβασμό 2,5 ετών. Ε, το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η αναθεώρηση αυτή θα έπρεπε να ε, συνδέεται με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ε, και τη διευκόλυνση του ε, διαλόγου του 2018, όπως επίσης και τον απολογισμό που θα γίνει από τις συνομιλίες του Παρισιού το 2023. Θα εξετάσει, θα υποβάλει τις τροπολογίες και θα συμμετέχει στην εξέταση αυτών με σκοπό την επικοδομητική συνεργασία. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γκούε, κύριε, κύριε Μπενίτο Σιλουάγκα, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σα Δεν θα σας ε, εκπλήξω αν σα πω ότι συμφωνήθηκε κάτι για την θερμοκρασία ε, ε, στο Παρίσι γιατί τη αυτή κατά πέντε βαθμούς είπαμε είναι φιλόδοξες οι, οι προτάσεις της Κομισιόν αλλά όχι αρκετά ε, γιατί εδώ μιλούμε για κάποιους τομείς που δεν καλύπτονται από το ETS ε άρα θα πρέπει να αποφύγουμε κάποια κενά τα οποία θα μας οδηγήσουν στο να μην τηρήσουμε τα συμπεφωνημένα. Επίσης δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι η οικονομία και το περιβάλλον είναι πράγματα τα οποία έρχονται σε σύγκρουση. Γιατί μπορούμε να ρυθμίσουμε ε, το θέμα ακριβώς όπως κάναμε και με την ε, ενεργειακή ε, αποτελεσματικότητα. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε με κάποιες προτάσεις το κείμενο της Επιτροπής. Αν η αφετηρία είναι το 2017, αυτό είναι κάτι το εύστοχο. Έτσι θα έχουμε εξοικονόμηση εκπομπών. Και επίσης θα είναι πιο εύκολο να προσαρμοστούν τα κράτη. Θα είναι πιο βαθμιαίο, πιο μαλακό, πιο εύκολο για να συμμορφούν τα κράτη με τους στόχους. Επίσης, ε, για τον έλεγχο συμφωνούμε, θα κατεβάσουμε και κάποιες τροπολογίες ε, σε σχέση με αυτή την αναθεώρηση που θα πρέπει να προσαρμοστεί ε, σε, σε όσα προβλήματα για, για το, Και επίσης θα πρέπει για τα κράτη-μέλη να ε, κάνουν κάποια προσπάθεια για αυτές τις προσαρμογές και αυτό να θεωρηθεί κάτι θετικό και όχι κάτι τιμωρητικό όπως συστήσαμε και χτες. Σε κάποια άλλα σημεία είμαστε κατά, εκεί δηλαδή που θεωρούμε ότι κάνουν πιο ε, δύσκολη τη διαχείριση της υπόθεσης αυτής. Αυτό πρόκειται να είναι κάτι ε, αυτά τα οποία προβλέπονται σε κάποια σημεία είναι κακά για τη γη. Δεν υπάρχει εδώ πέρα ξεκάθαρο χρηματοδοτικό πλαίσιο και θα πρέπει τι θα γίνει με τις αρνητικές εκπομπές και τη σχετική απορρόφηση. Όλα αυτά με κριτήριο τη συμμόρφωσή μας προς τις διεθνείς δεσμεύσεις. Ο κ. Σταμπουράνο είναι εδώ για το δηλαδή δεν έχει λόγο του το ε, ε, έχει ζητήσει το λόγο. Οπότε πάμε τώρα πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Μέτσκε που είναι ο Γενικός ε, Διευθυντής, τέλος που πρόκειται Γενική Διεύθυνση για το κλίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συμφωνώ με το Κοινοβούλιο ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια που καλύπτει το 60% των εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε από τώρα παρακαλώ να μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο παραπάνω από δύο λεπτά γιατί θέλω να σας πω τα εξής πέντε σημεία τα οποία έχουν σχέση με το σχέδιο γνωμοδότησης και σας ε, ευχαριστώ για το κείμενό σας. Πρώτα πρώτα όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη φιλοδοξία μας θα πρέπει εδώ πέρα να κάνουμε ε, κάποιο είδους διευκρίνηση τι εννοούμε γιατί έχει εδώ πέρα η πρόταση πρόκειται για κάποιες ε, ε, εκπομπέ για, για κτίρια, γεωργία, μεταφορέ Εκεί είπαμε ότι θα πρέπει να πάμε στο 0% μέχρι το 2040. Ε, πρώτα, πρώτα ε, διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν έχει περάσει από κάποια αξιολόγηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, οι συνέπειες εδώ είναι πάρα πολύ σκληρές, γιατί θα, πούμε, θα πρέπει να καταργήσουμε μέχρι το 2040 έγες, πρόβατα και αγελάδες. Μα είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο με το 2040. Καλά, να μην μπούμε για κτίρια και μεταφορές όσον αφορά το στόχο των, των μηδενικών του 2040. Επίσης, τι γίνεται με τις εκπομπές από την βιοενέργεια. Εδώ θα έχουμε με μεγάλη διαφορά και αλλαγή στο σύστημα που ισχύει τώρα όσον αφορά το ότι θα γίνει περίπλοκο το σύστημα έκθεση, ε, το σύστημα ε, της παγίδευσης Amendment number 10 is asking for is to account for under the non-ETS. Uh, it would also bring... Και με το ETS και εκτός του ETS γι' αυτό, για, για τη δέσμευση λέει, των εκπομπών. Άρα θα πρέπει η υποβολή της έκθεσης θα πρέπει να γίνεται διπλή η υποβολή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός άλλη έκθεση, άλλη αναφορά. Επομένως αυτό θα φέρει άχθος διοικητικότερο όσον αφορά αυτά τα credits για τη χρήση της γης. Δεν θέλω να σας πω τώρα για τα αριθμητικά δεδομένα, αλλά για το εύρος της εφαρμογής του μέτρου. Θα πρέπει εδώ να έχουμε κάποια συνέπεια. Να κοιτάξτε, ε, όσον αφορά τις εκπομπές από την εξαφάνιση των δασών. Αυτό πώς θα μετρήσει. Θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί. Αλλά και για την τροπολή 18 και 17, εκεί που έχει κάποια αριθμητικά στοιχεία, νομίζω ότι αυτά δεν... Κάτι, κάτι, κάτι, κάτι πάει στραβά, δεν ταιριάζουν τα, τα λοιπά. Τώρα όσον αφορά την συμμόρφωση, όντως εμείς προτείναμε έναν κύκλο πενταετή. Εάν πάμε σε μονοετή κύκλο συμμόρφωσης, τότε θα πρέπει να αλλάξει το πράγμα και για τη δασοπονία και για τη χρήση της γης, θα πρέπει δηλαδή να αλλάξει τρέχουσα πρακτική. Άρα να έχουμε αύξηση του δικαιωτικού άκθους για όλα τα κρατημέλη και σε βαθμό αρκετά αυξημένο. Έχει υπάρχει αυτή η πρόταση για τα 2,5 χρόνια να μην έχουμε επομένω αιτήσει υποβολή εκθέσεων, αλλά να έχουμε εξαμηνία για να καλύψουμε αυτά τα δυόμιση χρόνια. Και αυτό όμως θα είναι μεγάλη αύξηση του διοικητικού άρθρου, ούτως ώστε να εφαρμοστεί η πρόταση. Πέμπτον, έχουμε το άρθρο 10 και την τροπολογία 21. θα ήταν άδικη αυτή η ρύθμιση για τις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Πρόσοχη. Δεν θέλω να σταθώ τώρα στο θέμα της ευελιξίας, γιατί έχουμε την πρόταση για την ε, αφετηρία, ε, το ποσό κλπ. Εμείς έχουμε κάνει κάποια αξιολόγηση. Έτσι βέβαια θα ήταν ίσως πιο στεγνό το σύστημα, αλλά πρέπει να δούμε στην αξιολόγηση ποιες είναι οι συνέπειες. Τέλος, είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε γιατί τώρα να ξεκαθαριστεί η κατάσταση αλλά και όσον αφορά τις προτάσεις και τις επιπτώσεις αυτών. Επομένως θα συνεργαστούμε στενά τα μέσα εβδομάδες με τον εισηγητή αλλά και τους κοιόδης εισηγητές για την έκθεση της ΙΤΡΕ. Ε, Επιτροπή σας ευχαριστούμε. Τώρα, ας δευτερολογήσει ο κύριος Γιαβόρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και πολύ σύντομα θα ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης και την Επιτροπή για τις θέσεις τους, για τη συμβολή τους. Βεβαίως, διαπιστώνουμε κάποιες διαφορές τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ελπίζω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές θέσεις. Σημαντικό για μένα είναι να προχωρήσει ο κανονισμός και ε, με φιλοδοξίες σύμφωνες με τους γενικούς στόχους του περιορισμού των εκπομπών και της στήριξη των δεσμεύσεων των Παρισίων. Στα τεχνικά θα, θα βρούμε συμβαστικές λύσεις βεβαίως Λαμβάνω υπόψη και των προτάσεων των διαφορών εμπλεκομένων φορέων. Ευχαριστώ την Επιτροπή για τη διάθεση για περαιτέρω συζήτηση. Είμαι πεπισμένο ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση αποδεκτή για του πάντε. Ευχαριστώ κύριε Χαβόρ. 16 Ιανουαρίου, 6 το βράδυ, η προθεσμία για τις τροπολογίες, 30-31 Μαρτίου ψηφοφορία στην ΙΤΡΕ, 29 Μαΐου στην ΕΝΒΗ. Ολομέλεια ακόμα δεν έχει προσδοριστεί. Και ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση για να περάσουμε στο σημείο 9, αφού έχει αναβληθεί για τις 6 Φεβρουαρίου το σημείο περίθμων 8. 9. Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Συνεργατική Οικονομία. Γνωμοδότηση έχουμε υπό το άρθρο 54 του κανονισμού για την ΕΜΚΟ. Έχουμε αρμοδιότητα λοιπόν αποκλειστική σε ορισμένα ζητήματα. Συνδεδεμένη ψηφιακή οικονομία και νέε ευκαιρίε για τι επιχειρήσει και τον καταναλωτή, κυρίω μικρομεσαίες επιχειρήσει και πολύ μικρέ επιχειρήσει. Η καινοτομία ωστόσο αυτή αφήνει και αβεβαιότητε σε σχέση με τα δικαιώματα και τι δυνατότητε αυτή τη ψηφιακή οικονομία. Η ανακοίνωση της Επιτροπής στόχο έχει να δώσει απαντήσεις σε αυτές τις ανησυχίες και καθοδήγηση και βεβαιότητα ασφάλεια δικαίου για την αγορά, για τις επιχειρήσεις, για τους καταναλωτές. 30 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας για τη συζήτηση αυτή και δίνω το λόγο ξεκινώντας στον κύριο Ταμπουράνο ως εισηγητή από το EFTT έχετε το λόγο. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι και πρώτα απ' όλα καλή χρονιά Έχουμε ως καθήκον ε, να εκφράσουμε τις δικές μας προοπτικές για την συνεργατική οικονομία εμείς από την Επιτροπή μας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα γιατί έχουμε διαρκή εξέλιξη στον τομέα αυτών. Αφορά βέβαια και τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις μας, τους πολίτες μας και ε, όλους τους παράγοντες που βρίσκονται μεταξύ αυτών. Είτε πρόκειται λοιπόν για τοπική αυτοδιοίκηση, πόλεις, έθνη, κράτη ή με ευρύτερο επίπεδο έχουμε όλο και πιο συχνά την εισαγωγή της ψηφιακής οικονομίας και βέβαια πρέπει να εξασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ δύο παραγόντων. Καταρχάς την παρατήρηση και τη δημιουργία ενός παράγοντα ελευθερίας για την καινοτομία και την ε, τις δοκιμαστικές προσεγγίσεις και δεύτερον προστασία των εργαζομένων, των καταναλωτών, των παραγωγών ε, με βάση και βέβαια την αντίστοιχη προσαρμογή του διοικητικού μηχανισμού και της φορολογίας. Είναι σημαντικό εδώ να γνωρίζουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια πληθώρα μορφών συνεργασίας οι οποίες πάνε από την οικονομία της δωρεάς μέχρι την οικονομία που προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία της αγοράς και άρα πρέπει να μιλούμε για οικονομίες συνεργατικές, στον πληθυντικό δηλαδή και όχι για συνεργατική οικονομία. Βέβαια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μόνο διάστατη προσέγγιση. Not one size fits all, μας λέει η Επιτροπή. Και αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται η ποικιλία η πληθώρα που βρίσκεται στο τομέα αυτό. Πληθώρα βεβαίω με ελάχιστου κοινού παρανομαστές, μεταξύ των οποίων πρώτον ε, ο επιμερισμός ε, πόρων, είτε υλικών είτε Άιλον που σημαίνουν και οικονομία κοινωνική, περιβαλλοντική και αποτελεσματική ε, χρήση των πόρων, οικονομία κλίμακος, δεύτερον εμπλοκή ενεργός των ε, πολιτών, τρίτον υποδοχή της ε, συνεργατικής αυτής μορφής από την κοινότητα, γιατί οι κοινότητες αυτές που αποδέχονται τη συνεργατική οικονομία στηρίζονται στην, το μοίρασμα των πόρων και των γνώσεων, ανοίγουν open source, δημιουργούν νέα κοινά αγαθά, Creative Commons. Τέταρτον, έχουμε την εντατική χρήση των τεχνολογιών, της πληροφορίας, της επικοινωνίας και εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ε, ουσιοδέστατο παράγοντα και άξονα για ταχύτατη ανάπτυξη με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων ε, χάρη στους οποίους δημιουργείται το νέο προϊόν, η καινοτομία και βέβαια έχουμε χαμηλότερο άμεσο και έμεσο κόστος. Και έχουμε και την ε, διοχέτευση των πληροφοριών και την ενίσχυση βέβαια της ε, εμπιστοσύνης μεταξύ ισότιμων μερών. Έτσι λοιπόν πρέπει να επιδιώξουμε με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να ενισχύσουμε την απόδοση και την, το όφελος που προσφέρουν οι ε, συνεργατικές οικονομίες για τις επιχειρήσεις τους πολίτες, για τις κοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν μη αποκλειστικού χώρους δοκιμαστικής προσέγγισης των ε, συνεργατικών οικονομιών με ε, νομοθεσία ευνοϊκή προς αυτές σε ευρωπαϊκό, εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο, με ευνοϊκή προσέγγιση ως την, προς την ψηφιακή τεχνολογία και βέβαια την εισαγωγή της τεχνολογίας 3.0, της τρίτης εκδοχής δηλαδή του επίπεδου και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγυηθεί πως οι πολιτικές η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι συμβατές με το μέλλον και ότι θα προσφέρουν ασφάλεια δικαίου και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούμε να έχει αυστηρή στάση απέναντι στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους επιχειρηματίες, να εγγυάται την ασφάλεια για τον πελάτη, να εξασφαλίσει εργατικές δράσεις σε σχέση με παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, να βοηθήσει στον προσδιορισμό του, ε, και την περιγραφή της εργασίας και της παροχής υπηρεσιών ή της παρεχόμενης υπηρεσίας και εδώ σας περιγράφω μόνο κάποιες από τις ιδέες που έχω συζητήσει, ελπίζοντας ότι με τις προτάσεις και τις ε, τροπολογίες των συναδέλφων θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε με ε, σημεία και με διαστάσεις που δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να αναλυθούν με επάρκεια και βάθος. Αυτά και περιμένω να ακούσω τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ταμπουράνο. Δείξαμε ανοχή στην υπέρβαση χρόνου από πλευρά σας, γιατί δεν μιλήσατε καθόλου μέχρι τώρα και άρα λέμε ότι έτσι ισοσκελίζετε την μη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Ακούμε λοιπόν τους Σκιώδης με το ΕΛΚ πρώτο, η κυρία Σάντερ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή που ε, στη γνωμοδότηση του αναφέρεται στις διάφορες θεματικές ενότητες που έχουν να κάνουν με τη συνεργατική οικονομία. Αυτή την οικονομία ξέρουμε ότι έχει πολύ μεγάλο δυναμικό και έχει πολλά πλεονεκτήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πρωτοστατήσει στον τομέα αυτό. Δίνει τη δυνατότητα στους άνεργους, στους συνταξιούχους και στους νέους, στους φοιτητές και ενδεχομένως σε επισφαλώς απασχολούν να βρουν μια θέση απασχόλησης και να συμπληρώσουν ε, το εισόδημά τους. Ε, οι επιχειρηματίες θα ε, βρίσκουν καθημερινώς νέες υπηρεσίες και νομίζω ότι πρέπει να τους ενθαρρύνουμε και να συνοδεύσουμε την ανάπτυξη αυτών των νεοφιών επιχειρήσεων. Όσον αφορά το δίκαιο που ισχύει για ε, τους δημιουργούς και τους χρήστες αυτής της πλατφόρμας ε, ε, πρέπει να διευκρινιστεί. Το συνεργατική δεν πρέπει να αποτελεί μία επικάλυψη για αθέμητο ανταγωνισμό για τους τεχνίτες μας και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω κάποιες διευκρινήσεις και προτάσεις που θα αφορούν κυρίως τη σημασία των, του αθέμητου ανταγωνισμού, όπως επίσης και την ύπαρξη και ε, απόκτηση δεξιοτήτων ε, ε, από τους χρήστες, όπως επίσης και τη δυνατότητα πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω της πλατφόρμας. Η συνεργατική οικονομία βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Προτείνω λοιπόν την ανάπτυξη μηχανισμών πιστοποίησης ε, των ε, απόψεων των καταναλωτών, ώστε να ε, μην υπάρχει πληθώρα κακών ε, γνωμοδοτήσεων, ε, όπως τις αποκαλούμε. Πρέπει να έχουμε ε, πλήρη και ακριβή δεδομένα. Πρέπει συνεπώς να ενισχύσουμε ε, την ύπαρξη μηχανισμών που μπορούν να διακρίνουν ε, τις ε, αμοιβόμενες από τις μη αμοιβόμενες δραστηριότητες μεταξύ άλλων και πρέπει να ενημερώνονται οι χρήστες για τους ισχύοντες κανόνες και να γίνεται καλύτερος έλεγχος του σεβασμού της νομοθεσίας. Εν τέλει κύριε Πρόεδρε έχω ένα ερώτημα σε σχέση τη διαδικασία και θα ήθελα επειδή την επόμενη εβδομάδα θα, ε, ε, θα έρθετε στο Στρασβούργο, ε, θα είστε στο δρόμο, μήπως θα μπορούσαμε να καθυστερήσουμε κατά μία μέρα της την προθεσμία υποβολής τροπολογιών και να την μεταφέρουμε την Τρίτη αντί για τη Δευτέρα. Ναι, νομίζω 3η 17 Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι έχει είναι πλέον η νέα μας ε, προθεσμία, οπότε αυτό έχει ε, καλυφθεί. Θα το έλεγα στο τέλος της συνεδρίασης. Ε, οι σοσιαλδημοκράτες εκπροσωπούνται σήμερα από την κυρία Ντεμόντε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για το κείμενό του. Το κείμενό του είναι σύντομο αλλά αυτό Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε το πόσο σημαντική είναι η συνεργατική οικονομία. Ε, όλο ένα και πιο σημαντική είναι για την οικονομική δραστηριότητα που αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πρόκειται για ένα νέο μοντέλο. Για δυσκολία θα πρέπει να δούμε πώς θα το ε, ρυθμίσουμε, ε, γιατί θα γίνει στο μέλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί, πιο αποφασιστικοί στο κείμενο για νέες στρατηγικές και πολιτικές. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με σύντομη προθεσμία που έχουμε για κάποιες ε, τροπολογίες. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, εγγύησεις υπέρ των προσωπικών δεδομένων, να υπάρχει ομοιογένεια, να υπάρχει συνοχή μεταξύ του τι κάνει το κάθε κράτος ε, μέλος επιμέρους για να δούμε τι θα γίνει με την ε, κάθε εθνική νομοθεσία, αλλά να δούμε και τι ενέργειες θα ε, αναλυφθούν τοπικά και περιφερειακά. Γιατί έχουμε πολλά είδη πλατφόρμας ε, για την ευελιξία, για την κινητικότητα των εμπλεκομένων. Όλα αυτά θα πρέπει να οριστούν με προσοχή. Να μην υπάρχει δυνατότητα μονοπωλίου για αυτές τις πλατφόρμες. Βέβαια αυτό είναι θέμα εσωτερικής αγοράς και ανταγωνισμού, αλλά το τονίζουμε και εν προκειμένου. Όταν θα γίνει με τους ε, παρόχους υπηρεσιών και εκεί θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη ε, ρύθμιση. Ε, επίσης να δούμε τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις που δίνουν σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει και εδώ να υπάρχει ξεκάθαρο φορολογικό πλαίσιο και να υπάρχει και ευκολία πρόσβαση στην ταινιοδότηση. Εδώ πρόκειται για ανεξάρτητη ελευθέρεια τέλο πάντων, ελευθέρεια επαγγέλματα για αυτούς τους τομείς. Άρα θα πρέπει ένας ανεξάρτητος φορέας να διαχειρίζεται αυτό το τομέα με καθημερινές γραμμές, και να είναι κοντά στους εμπλεγωμένους. Οι περιφερειακές περιοχές είναι κάτι που βρίσκει σύμφωνο, γιατί και στην Επιτροπή των μεταφρών. είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση μεταξύ των μεγάλων πόλεων και των άλλων. Υπότιτλοι για σημαντικές ε, υπηρεσίες ακριβώς που έχουν σημασία για τις πιο ορεινές περιοχές. Εν κατακλείδη έχουμε και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Εδώ προσοχή επισχή, επικουρικότητα και για αυτήν την στρατηγική. Ευχαριστώ ε, κύριε Αντεμόντη. Κύριος Χένκελ δεν μπορεί να είναι εδώ. Όμως ο κ. Τουρσινόφσκι θα τον ε, εκπροσωπήσει εκ μέρους της ECR. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, ζήτησω συγγνώμη εκ μέρους του σκιώδου συζητητή μας, ε, τον αντικαθιστό. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσει τον εισηγητή θεωρεί ότι μια συνεργατική οικονομία είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να ε, είναι ε, μικρότερο το κόστος των υπηρεσιών για τους ε, χρήστες και επίση είναι και πιο ευέλικτες οι ευκαιρίες απασχόλησης που θα προκύψουν. Μπορούμε να προωθήσουμε την ψηφιακή αγορά, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να είμαστε κατά των πλατφορμών ε, οπότε επικροτούμε την ε, προσέγγιση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν ειδικοί φορολογικοί κανόνες, ειδικότερα για τις υπηρεσίες εστίασης, για παράδειγμα, που πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές όσον αφορά την υγιεινή και όσον αφορά όσους απασχολούνται στον τομέα των μεταφορών πρέπει επίσης να πληρούν κάποιους ε, όρους και προϋποθέσεις ειδικού. Ε, η συνεργατική οικονομία μπορεί να βελτιώσει επίσης την ποιότητα των υπηρεσιών ε, και να παίξει το ρόλο της ρύθμισης σε, παραδοσιακέ σε παραδοσιακές δομές. Αναφέρομαι περισσότερο στα φορολογικά συστήματα γιατί μπορεί να υπάρχουν ε, ιδιαίτεροι κίνδυνοι στο πλαίσιο της συνεργατικής ε, οικονομίας ε, και πρέπει να βοηθήσει και η συνεργατική οικονομία στην, ενίσχυση της, μείωση τη της της Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας και ε, εντός χρόνου. Ο κύριος Ρίκη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ταμπουράνο που ε, υπόσχεται πολλά και είναι και ε, πολύ σύντομη η έκθεση. το πρόβλημα της συνεργατικής οικονομίας είναι ότι έχει τρία σκέλη. Πρώτον, ένας προμηθευτής, ένας πάροχος που μπορεί οτιδήποτε να προμηθεύσει ως ε, υπηρεσία ή αγαθό, από την άλλη ένας ε, πελάτης, ε, καταναλωτής, ο οποίος είναι ο αποδέκτης και διαμέσως μία πλατφόρμα ψηφιακή που διέπεται από περίπλοκες αρχές και το πρόβλημα είναι ότι η ψηφιακή οικονομία πρέπει να συνδέεται με το υπόλοιπο της οικονομίας. Συνεπώς πρέπει να δούμε πώς θα το οργανώσουμε, να προβληματιστούμε και πώς θα το ρυθμίσουμε όλο αυτό. Ολόκληρη την οικονομία σε όλο της το φάσμα ε, πηγαίνει κάπως προς όλες τις κατευθύνσεις ε, γιατί ε, ανάλογα με τις διαθέσεις του καθενός ο καθένας μας τα επιμείνει σε διαφορετικά σημεία. όμω υπάρχει ένα κοινό μα σημείο που είναι η προστασία των καταναλωτών, η προστασία των εργαζομένων, όπω επίση και την ποιότητα των δεδομένων. Νομίζω ότι η πραγματική δυσκολία λοιπόν είναι η... να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, να είναι μια οικονομία που θα καλύπτει όλο το φάσμα τη οικονομία. Ε, η ρυθμίση για την ώρα δεν είναι επαρκή και είναι και πολύ διασκορπισμένη. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να αρχίσουν να προβληματίζονται και να ρυθμίζουν την όλη διαδικασία. Πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ της συνεργατικής ε, εμπορικής οικονομίας, της αγοράς δηλαδή, και της μη κερδοσκοπικής, γιατί δεν πρόκειται καθόλου για την ίδια κατηγορία υπηρεσιών και πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένοι ε, ορισμοί για τη διάκριση αυτών ε, των δύο ειδών. Επίσης, αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι, ότι πρέπει να προστατεύσουμε και ε, τους πελάτες, τα δικαιώματά τους, τα, ε, δεδομένα τους, τους εργαζομένους, τα κοινωνικά τους δικαιώματα, τις ε, συμβατικές τους ικανότητες, ε, την αμοιβή τους κλπ πρέπει να ρυθμίσουμε τις πλατφόρμες ε, και σε φορολογικό και σε κοινωνικό επίπεδο και θα πρέπει επίσης ε, να εξετάσουμε μία ομογενοποίηση σε επίπεδο ευρωπαϊκό τουλάχιστον όσον αφορά τις, ε, τους γενικούς κανόνες και τη φορολογία ώστε όλη η κοινωνία να βρίσκεται σε μία, περίπου παρόμοια, σε μία παρόμοια θέση. Νομίζω λοιπόν ότι ο ορισμός Τη ε, της ε, ρύθμισης είναι πάρα πολύ σημαντικός και έχουμε τεράστια δουλειά να κάνουμε ε, στο πλαίσιο όλων των οργάνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρικέ. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπες από τους Σοσιαλιστές θέλει να πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις προτάσεις του κειμένου του. Ε, βέβαια, και τώρα έχουμε αυτή και μεγάλη αλλαγή του κοινωνικού μοντέλου και της οικονομίας για αγαθά και υπηρεσίες. Έτσι θα στηριχτεί η οικονομία μας. Αλλά αυτό θα ε, σημαίνει και για το πώς κινούμεθα, πώς ταξιδεύουμε, τι εργασιακές σχέσεις θα υπάρχουν. Θα πρέπει να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν μέχρι να υποβληθεί αυτό το σχέδιο. Πάντως θα κατεβάσω κάποιες τροπολογίες ούτως ώστε να δείξω κάποια συγκεκριμένα ζητήματα αυτού αυτό το κείμενο ακριβώ όπως τις υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ειδών πλατφόρμας. Γιατί θα πρέπει να το θα κάνουμε με τις αλλαγές σε εργασιακές σχέσεις, γιατί τι θα γίνει με τα μονοπόλια που αυξάνονται και επίσης για τη φορητότητα ε, όσον αφορά τα ψηφιακά της κάθε πλατφόρμας. Ευχαριστούμε κύριε Μπλάνκο Λόπες. Δεν ζήτησε άλλο το λόγο. Άρα πάμε στον κύριο Νίλκε, ήμουν εκπρόσωπο τη ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, ε, αρμόδια γενική διεύθυνση. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Το κοινοβούλιο για την γνωμοδότηση. Πού αφορά την ανακοίνωσή μα. Πάρα πολύ αυτά όσα παρατηρήσατε. Εγώ θα σταθώ σε κάποια από αυτά που αναφέρατε πρώτα πρώτα. Το θέμα με αυτήν την εργατική οικονομία είναι το ότι διακρίνεται από πολυμορφία. Πλατφόρμες, παρόχους, ε, καταναλωτές, πελάτες. Οπότε θα πρέπει εδώ να γίνει διαχωρισμός. Όπως είπαμε ότι υπάρχει διαφορά ε, όσον αφορά κάποια υπηρεσία που παρέχει μία επιχείρηση. Και εδώ είναι θέμα επίσης και ε, νομοθεσίας. Τι γίνεται λοιπόν με αυτούς τους παρόχους της πλατφόρμας. Και γι' αυτό η ανακοίνωσή μας διακρίνεται από κάποια ε, επιφυλακτικότητα όσον αφορά νέα νομοθεσία. Ή ένα νέο κανονισμό γιατί ακόμα υπάρχουν κάποιες φεζόνες για αυτές τις υπηρεσίες των πλατφορμών. Νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Ότι δηλαδή παρά το ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε τα πλεονεκτήματα της συνεργατικής οικονομίας για την απασχόληση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε δίκες συνθήκες ανταγωνισμού, να κατοχυρωθούν, να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και των καταναλωτών. Δηλαδή να καταλήξουμε σε κάποιο σχήμα που να είναι ωφέλιμο για όλους. Εμείς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Πρόκειται για κάποιους τομείς που εξελίσσονται πολύ γρήγορα πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη οικονομία και την ανάπτυξή της. Και το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Οπότε συμφωνούμε μαζί σας και θα ξεκινήσουμε δύο συμβάσεις εποπτείας παρακολούθησης, ούτως ώστε να καταλάβουμε καλύτερα ποιες είναι οι επιπτώσεις της νέας αυτής νομοθεσίας για την οικονομία. Και να δούμε τι θα γίνει από πλευράς ανάπτυξης οικονομίας και το τι είδους ανάπτυξη θα προκύψει. Άρα θα σας ενημερώνουμε και θα σας ε, λέμε το πώς θα εξελιχθεί η δουλειά μας στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πρόεδρος εδώ ολοκληρώνεται αυτό το θέμα, αλλά πρώτα θα πρέπει να δευτερολογήσει ο κύριος Ταμπουράνο, εισήγητης. Είμαι πολύ σύντομος, ε, γιατί όσο παρουσίασε την έκθεση, εξήνισε το χρόνο, στο όλους έλαβα το λόγο. Ναι, θα πάρα πολύ καλά θα τα πάμε και το σαν Ντάντι θα κάνουμε ότι γίνεται καλύτερο. Ο Πρόεδρος, ε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ταμπορανό. Και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό. Και περνούμε στις ανακοινώσεις για το χρονοδιάγραμμα ως συνήθως, όπως είπε και η κυρία τροπολογίες. 16, από 16 Ιανουαρίου στις 6 πάμε στις 17, Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι. Τρίτη 17 στις 12 το μεσημέρι, έχετε μερικές ώρες παραπάνω στη θέσή σας. Ψηφοφορία στην Ήτρε στις 28 Φεβρουαρίου, στην Καθήλυνα Αρμόδια ΙΜΚΟ 24 Απριλίου και ολομέλεια ακόμα δεν έχουμε προσδιορίσει. Και περνώ στο σημείο 10 στην ημερήσια διάταξη, ενημέρωση σχετικά με τι ανεξελίξει διαπραγματεύσει. Το φάσμα πρώτα, μετά η περιαγωγή χονδρική και εν τέλει το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών. Θα κάνει παρουσίαση ο κάθε εισηγητή κάθε φορά και αν περισσεύει χρόνο. θα αφήσουμε και του συναδέλφου. Βέβαια χρόνο όπω βλέπετε έχουμε, οπότε υπάρχει περιθώριο για συζήτηση με το πρώτο θέμα λοιπόν, το φάσμα. Κυρία Πατρίτσια Τόγια είναι η εισηγήτρια για τη σχετική απόφαση. 13 Δεκεμβρίου έλαβε χώρα ο πρώτος τριμερής διάλογος. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Τόγια λοιπόν και να δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Ωστόσο είναι σε άλλη συνεδρίαση. Θα διαπιστώσατε στην ψηφοφορία ότι ήταν κάπως βιαστική. Την αντικαθιστά όμως η κυρία Κομπλανάντρη που θα μας ενημερώσει εκ μέρους της παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε και θα μεταφέρω τους χαιρετισμού του Προέδρου και στην κυρία Τόγια και τα συγχαρητήρια. Ήτανε ε, αναπάντηχο το ότι επέτυχαν τόσο γρήγορα μια συμφωνία. Ίσως το πνεύμα του Χριστουγέννων έφτασε και μέχρι το Στρασβούργο. Έφτασαν λοιπόν σε συμφωνία. Εγώ πριν από πολύ λίγα λεπτά έλαβα τη σχετική, ε, το σχετικό σημείο από την κυρία Τόγια και έτσι αν υπάρχει συνάδελφος που ήταν στον τριμερή διάλογο, ας λάβει το λόγο παρακαλώ. Εγώ έχω ένα υπόμνημα μόνο από το γραφείο της κυρία Στόγια. Λοιπόν, έγινε η τεχνική συνεδρίαση για να προσδιοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες. Από ό,τι βλέπω, με χαρά διαπιστώνω ότι είναι καλό το κείμενο, με δεκτές τις προτάσεις και τι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αποτελεσματικότητα του φάσματος. Γενικά είναι ικανοποιημένη για την τελική συμφωνία που υλοποιεί και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιμένουν από το Κορεπέρ ε, τις θέσεις και την έγκριση από τα κράτη-μέλη. Αυτές τις μέρες αναμένεται με 26 ε, του μηνός χρονοδιάγραμμα κατά πάσα πιθανότητα και βέβαια μετά πάει στην Ολομέλεια. Κάποια σημεία που έχει λόγο να αναφέρουμε. Για δύο χρόνια, ανάλογα βέβαια με την αιτιολόγηση που μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο ειδικό παράρτημα παραμένουν τα 100 MHz ως στόχος, ως παρατείνεται δηλαδή, αλλά βέβαια πρέπει να ευθυγραμμίζονται στους στόχους ε, που έχουν αναφερθεί στο πρόγραμμα για το φάσμα τα κρατημέλη, για τα 700 MHz έως το 2030 τουλάχιστον θα έχουν φέρει αυτή την ευρύτητα, τα κρατη από την άλλη διαφορές μεταξύ πλατφόρμας, ίντερνετ και άλλων υπηρεσιών διαγράφεται. Και διαγράφεται επίσης και η αναφορά στο downlink, δηλαδή δεν ισχύει μόνο για το κατέβασμα αλλά και για το ανέβασμα περιεχομένου. Άρα έχουμε ισότιμη μεταχείριση όλων των εμπλεκομένων. Το 5α έχει μεγάλη σημασία ως άρθρο γιατί εδώ τα κράτη-μέλη ε, εισάγουν κανόνες για να περιορίσουν υπέρ του καταναλωτή τις συνέπειες ε, της, ε, των κλειδονισμών που μπορεί να σημάνουν αυτές οι νέες τεχνολογίες και η αξιοποίηση βέβαια του φάσματο στα 700 MHz θα έχει πολύ μεγάλη σημασία κτλ. Πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τρόπο σωτμίο για να προωθηθούν όλα τα θέματα τα πολιτιστικά. Ευχαριστώ. αυτέ ήταν οι πιο σημαντικέ παρατηρήσεις. Από ό,τι βλέπω δεν ζητεί κανεί άλλο το λόγο. Και συγχαίρω τη συνάδελφο για την τόσο αποτελεσματική ενημέρωση. Ευχαριστούμε και εμείς και συγχαρητήρια στην κυρία Τόγια. Και Περνούμε στην ενημέρωση για τον άτυπο διάλογο για την περιαγωγή με εισηγήτρια την κυρία Κουμπλανάτρη εκ μέρους Επιτροπής μας. Πρώτος τριμερής για τις 14 Ιανουαρίου, ο προσεχής προγραμματίζεται στις 7 Φεβρουαρίου. λυπούμε, ξέχασα να πω ότι 26 Ιανουαρίου θα γίνει ψηφοφορία για το φάσμα. Ε, επανέρχομαι στην περιαγωγή. Ο τριμερής λοιπόν, ο δεύτερος ε, προβλέπεται για τις 17 Ιανουαρίου και περιμένουμε να δούμε και εκεί ε, εξελίξεις. Κυρία Κουμπλανάτρη πάλι για πέντε λεπτά θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζομαι πέντε λεπτά επειδή είχαμε μια πολύ καλή αρχή ε, στην Επιτροπή μας με όλους και όλους ε, εισηγητές. Θα είναι πολύ μεγάλη υποστήριξη για την ε, γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μόνο έναν τριμερή διάλογο είχαμε πριν από το φάσμα Στι 14 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο και ο επόμενος ε, τριμερής διάλογος, ε, επειδή εγώ θα ήθελα να πάμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να είμαστε έτοιμοι για την περιαγωγή για τους χρήστε στην Ευρώπη μέχρι τον Ιούνιο του 2017, όμω, ε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Το να έχουμε από απόψε καθαρά είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδύνατο σχεδόν να έχουμε για την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ε, αίθουσα. Αν τα καταφέρουμε θα είναι Τετάρτη, 8 η ώρα το βράδυ. Ε, Θέλουμε να είναι έτοιμοι οι τριμερείς διάλογοι μέχρι τις αρχές ε, Φεβρουαρίου για να μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που έχουν, έχει τεθεί. Θέλουμε να τελειώσει αυτό το θέμα της περιαγωγής. Όλες οι πολιτικές ομάδες το θέλουν αυτό. Ε, επειδή έχουμε παρακολουθήσει την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου, εγώ θα ήθελα να πω ότι το Συμβούλιο είχε μία πολύ αδύναμη πλειοψηφία, με το ζόρι πλειοψηφία πλειοψηφία, ενώ στο Κοινοβούλιο ήταν πολύ πιο ε, μεγάλη η πλειοψηφία. Οι βασικές διαφορές αφορά τις τιμές ε, των δεδομένων, ε, της επικοινωνίας και γενικότερα το τίμημα που πρέπει να πληρώσουν μεταξύ τους πλέον οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών και εφόσον οι χρήστες δεν το πληρώνουν πια. Ελπίζουμε μέχρι μέχρι τον επόμενο τριμερή διάλογο, επειδή υπήρξε και κάποια διαβούλευση με τους χρήστες τα τέλη του 2016, ελπίζω να είμαστε έτοιμοι μέχρι τον επόμενο τριμερή διάλογο. Ελπίζουμε να έχουμε ε, ε, χρήση απεριόριστη των δεδομένων, ε, να τελειώσει η περιαγωγή, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι προορισμοί για τους χρήστες, ενδεχομένως ότι δεν μπορεί κανείς να έχει 300 GB ε, και να, τη στιγμή που ταξιδεύει για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για τους καταναλωτές οι τιμές ε, τώρα, ε, ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τις ε, πλέον πρόσφατες πληροφορίες και εμείς έχουμε κάποιες πληροφορίες και τεχνικές λεπτομέρειες εν ώψη των τριμερών διαλόγων την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω ότι θα έχουμε και στη διάθεσή μας μέχρι τότε από πολιτικής απόψεως τα στοιχεία που χρειαζόμαστε, τι ακριβώς θέλουμε να επιτύχουμε. Πρόκειται για ιδιωτικέ εταιρείε, είναι μια ε, ιδιωτική αγορά και προσπαθούμε να ρυθμίσουμε κάτι σε επίπεδο χονδρικής, οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Θέλουμε πάντω ε, να είμαστε ε, έτοιμοι και να θέσουμε τη βάση για τις ε, εσωτερικές ε, αγορές ε, που θα είναι πιο φιλικές προς τους καταναλωτές. Βρισκόμαστε να γνωρίζουν, να αισθάνονται ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αυτό έχει μία, έναν αντίκτυπο καθημερινό ε, και ότι δεν χρειάζεται κανείς να πληρώνει περισσότερο όταν αλλάζει ε, πάροχο τηλεφωνίας, ε, όταν μεταβαίνει από τη μία χώρα στην άλλη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ξέρω ότι ο κύριος Τροσανόφσκι είναι σκιώδης εισηγητής και εκείνος. Θέλετε να πάρετε το λόγο, κανείς άλλος δεν έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Ε, η ε, συγγήτρια παρουσίασε τον πρώτο τριμερή διάλογο ε, πολύ καλά. Τώρα το θέμα επαφίεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη ρύθμιση του θέματος των δεδομένων. Θα ήθελα να πω ότι είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Ε, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, να συγχαρώ πάντως την ησυχήτρια, γιατί είναι δύσκολο το θέμα. Πλησιάζουμε στο, στην εκπνοή της προθεσμίας οπότε ελπίζουμε να ε, έχουμε προχωρήσει. Βεβαίως πολλά εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε όμως ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τους διαλόγους πολύ σύντομα γιατί Έχουμε πραγματικά την προθεσμία ολόκληρου αυτού του εγχειρήματο και θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, κύριε Τοσενόφσκι. όπω είπε και η εισηγήτρια, η επόμενη συνεδρίαση προβλέπεται για τις 17 Ιανουαρίου και η κυρία Κομπουλανάτρη θα, θα ε, μας ενημερώσει 18 ε, Ιανουαρίου διορθώνει ο Πρόεδρος. Ε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όλες αυτές τις προσπάθειες, αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και ε, για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή μας. Πολλές πολιτικές ομάδες υποστηρίζουν αυτές τις πολιτικές απόψεις. Ε, πραγματικά σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Τετάρτη βράδυ θα αργήσετε να κοιμηθείτε. Πάμε τώρα ε, στο θέμα του συστήματος ε, εμπορίας εκπομπών αερίων, ε, για το οποίο θα κάνω την παρουσίαση εγώ και θα πρέπει τώρα εγώ να τηρήσω τα τρία λεπτά. Α, πέντε, πέντε, αλλά δεν θα χρειαστώ πέντε λεπτά. Λοιπόν, η γνωμοδότηση για το θέμα αυτό της Επιτροπής μας ψηφίστηκε στις 18 Οκτωβρίου, εγκρίθηκε από τη νομική υπηρεσία. Η θετική έκβαση της νομοδοσίας δίνει στον εισηγητή σαφή εντολή να εκπροσωπήσει την Επιτροπή μας στις διαπραγματεύσεις. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα να έχω μια εξισορροπημένη έκθεση που στέλνει ένα ισχυρό ε, μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στους εμπλεκόμενου φορείς ε, του συστήματος ε, εμπορίας ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να συνεργαστούμε στο πλαίσιο ενός μεγάλου συμβιβαστικού πακέτου και θα θυμάστε ότι ήταν σύντομη ψηφοφορία για το θέμα αυτό, γιατί ε, το ΕΛΚ, οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι συντάχθηκαν με την ε, βασική θέση της πλειοψηφίας ε, και οι υπόλοιπε ομάδες συμφώνησαν με κάποια σημεία του συμβιβασμού. Επίσης ε, έγιναν διαπραγματεύσεις και στην ΕΜΒΗ και είδαν με πολύ όρεξη ε, όλα όσα κάναμε εμείς στην Επιτροπή μας. Κάποια σημεία λοιπόν ε, ελήφθησαν υπόψη και φάνηκε αυτό και στην ψηφοφορία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Όσον αφορά τα διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης και αυτό αντανακλάται στην έκθεση Επιτροπής Περιβάλλοντος σημαντικά θέματα και σε συμβολικό επίπεδο αλλά και σε αριθμητικό επίπεδο είναι το θέμα της δημοπράτησης, ε, η ισορροπία ε, πλησιάζει πολύ στη δική μας άποψη και στα αποτέλεσμα της δικής μας ε, ψηφοφορίας όσον αφορά την διαρροή ε, άνθρακα ε, και εκεί τα καταφέραμε πολύ καλά όσον αφορά το έμεσο σύστημα αποζημίωσης και αυτό ε, εμφανίζεται στην έκθεση της ΕΝΒΗ. Υπάρχει μια σαφή συνοχή μεταξύ του καταποκοπήν ε, ορίου, το οποίο είχαμε προτείνει εμείς και συμφώνησε και η Επιτροπή Έμβη. Όσον αφορά τώρα τις κοινέ αρμοδιότητες, θα έλεγα ότι είμαι περήφανος ε, για μας και για το ότι καταφέραμε να περάσουμε τις απόψεις μας. Για μένα ο στόχος ήταν ε, να επιστρέψω εδώ με ένα κείμενο που μπορούμε να υποστηρίξουμε και στις διαπραγματεύσεις αλλά και στο πλαίσιο της Επιτροπής και πράγματι ε, υπήρξε συμφωνία, κατά τις τελευταίες ημέρες φαινόταν δύσκολη συμφωνία αλλά τελικά τα καταφέραμε, υπάρχει συμφωνία και εν ώψη του νέου πακέτου που ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση ε, επικαλυπτόμενων πολιτικών ε, να έχουμε ενεργειακά πακέτα το θέμα της συστήματος, του συστήματος ε, ε, εκπομπών αερίων και άλλα θέματα παράλληλα ε, πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν χρειάζεται να υπολογίζουμε τα ίδια δεδομένα πολλές φορές εντός των διαφόρων προγραμμάτων γιατί αυτό είναι επιπλέον άχθος για τον τομέα. Έχουμε επίσης ασκήσει πιέσει στο Συμβούλιο να ξεπεράσει το αδιέξοδο αλλά θέλουμε και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στον τομέα οι σκιώδη οι συζητητές ε, ε, θα προσπαθήσουν ε, σε συνεργασία μαζί μου κατά τις επόμενες εβδομάδες. Θα προσπαθήσουμε την επόμενη εβδομάδα να βρούμε λίγο χρόνο να, να συναντηθούμε για να το συζητήσουμε να δούμε κατά πόσο υπάρχει συμφέρον να επανυποβάλλουμε κάποιες ε, τροπολογίες. Ε, θα δούμε. Δεν ξέρω ακόμη τι θα γίνει. Θα το συζητήσω και με τους συναδέλφους. Αυτά από μένα όσον αφορά το σύστημα εκπομπών αερίων. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο? Ναι, Κύριε Μπούζεκ, ξέρουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θα ήθελα εσάς ε, να σας συγχαρώ ως εισηγητή ε, εκ μέρους της Επιτροπής Ήτρη. Ήταν πολύ σημαντική η γνωμοδότησή μας και ήταν πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος επί τη βάση του κανόνα 54. Δεν ήταν εύκολο να ε, το επιτύχουμε αυτό γιατί την τελευταία φορά στο σύστημα εκπομπών αερίων ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και εμείς δεν συμμετείχαμε καθόλου. Είναι μεγάλη ευθύνη και για τη δική μας την Επιτροπή και έχουμε και μεγάλη ευθύνη ενώπιον ε, της βιομηχανικής μας κοινότητας, επιχειρηματική μας κοινότητας, ε, του ενεργειακού τομέα και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την συνεργασία σας με την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Ήταν πάρα πολύ καλή και τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ε, όχι ε, μόνο εντός της ε, επιτροπής μας. Ε, νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να επανυποβληθούν κάποιες τροπολογίες γιατί υποστηρίχθηκαν από τεράστια πλειοψηφία στην επιτροπή μας. 85% των μελών της Επιτροπής μας υποστήριξαν τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Επίσης υπήρχαν συμβιβαστικές τροπολογίες που αφορούν την πραγματική μας οικονομία. Θα θέλαμε να εκπληρώσουμε όλες τις προδοκίες που αφορούν τη Συμφωνία του Παρισιού. Θέλουμε να έχουμε μία ε, βασική τοποθέτηση ε, ηγετική, ε, όμως ε, δεν θέλουμε να ε, σκοτώσουμε τη συμφωνία του Παρισιού και πιστεύω ότι θα είναι σημαντικό αν μπορέσετε να επανυποβάλλετε κάποιε από αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούζεκ, λέει ο Πρόεδρος, θα επανέλθουμε για το ζήτημα αυτό και εγώ έχω διαβουλευτεί με τους συναδέλφους. Είναι πάντως μια δυνατότητα, κύριε Μπούζεκ. Ο κύριος Τοσενόφσκι έχει ζητήσει το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Τοσενόφσκι. Eh, eh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω τις θέσεις της ομάδας του ECR. Εκφράζω στην ικανοποίησή μου για τις προσπάθειες που ξέρω ότι καταβλήθηκαν. Πολλά είναι τα κενά, ξέρουμε. Και είναι δύσκολο να βρούμε καλές συμβαστικές λύσεις και γι' αυτό θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Ένβη έλαβε υπόψη της, τη δική μας νομοδότηση. Και επαναλαμβάνω τα λόγια του κυρίου Μπούζεκ. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω στην τελική φάση αυτής της δουλειάς να συγχωνευθούν ή να ενοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο οι γνωμοδοτήσεις ΕΝΒΙ και ΙΤΡΕ. Γιατί ήταν ε, με όλο το γεγονός ότι εγκρίθηκαν δύσκολο να βρεθούν οι συμβαστικές ε, λύσεις. Άρα ελπίζουμε και δικές μας νομοδοτήσεις να εμφανιστούν στους τελικούς καταλόγους ψηφοφορίας σας. Και βεβαίως θα υποστηρίξουμε την έκθεση στην Ολομέλεια. Έχει μεγάλη σημασία όμως να μην λησμονήσουμε και τα συμφέροντα της βιομηχανίας, γιατί μερικές φορές φαίνεται να μην λαμβάνονται υπόψη επαρκώς Αλλά όπως είπα, είναι πάντα ευπρόζεκτη η συνεργασία μεταξύ ΕΝΒΙ και Ήτρε, γιατί δεν την είχαμε πάντα δεδομένη στο παρελθόν. Ο πρόεδρος ευχαριστώ πολύ. Σαφές το μήνυμα προς τους Κιώδης. Φαντάζομαι και οι απόντες αυτή τη στιγμή θα ενημερωθούν. Την επόμενη εβδομάδα σε όλους με τις διαβουλεύσεις θα γύρω και εγώ το θέμα. Εκ μέρους και του κυρίου Μπούζε και του κυρίου Τουσινόφσκη. Πάντως είμαστε σε μια καλή γραμμή. Πολλά από τα θέματα που μας έχουν αναφερθεί δείχνουν πρόοδο. Ο κύριος Μπούζακ είπε ότι η Ήτρε είχε 80% υποστήριξη. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντα βέβαια πρέπει να υποχωρούμε και να κάνουμε παραχωρήσεις, αλλά Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και με το τελικό αποτέλεσμα. Δεν βλέπω άλλη παρατήρηση στο θέμα αυτό. Άρα κλείνω το σημείο αυτό. Πηγαίνω στο 11, στα διάφορα. Δεν ζητεί κανεί το λόγο και πάω στι προσεχείς συνεδριάσεις 25-26 Ιανουαρίου του 2017 από τι 9 έως τι 12.30 και από τι 3 έω τις 6.30 στις Βρυξέλλες. Σας εύχομαι και πάλι καλή χρονιά και ευχαριστώ για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.